Άρχεται η συνεδρίαση της Ολομαλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνέχεια μετά από τη διακοπή της 9 η Ιουνίου του 2011. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 9 η Ιουνίου και τα κείμενα τα οποία ενεκρίτησαν σας έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις? Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά.